Ε, και της δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μογκυρίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. We face the biggest humanitarian... Είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση, τραγωδία στην περιοχή μας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. 6,5 εκατομμύρια Σύριοι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι και αν συνεχίσουν ε, οι εχθροπραξίες, αυτοί μπορεί να είναι οι αυριανοί πρόσφυγες. 400.000 περίπου Σύριοι δεν έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι υποπολιορκία. 4,6 εκατομμύρια είναι πλέον οι Σύριοι πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες με μεγάλες πιθανότητες να συνεχίσει να αυξάνεται αυτός ο αριθμός λόγω των έντονων σειράξεων και των μαχών ε, στο έδαφος. Ο λιμός στη Συρία χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο κατά των ε, πιο ευάλωτων, κυρίως γυναικοπαίδων, που λιμοκτονούν κυριολεκτικά. Η Συριακή κυβέρνηση τώρα έχει εξασφαλίσει ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ε, ε, αλλά δεν ε, αρκεί αυτό. Και σε άλλες πόλεις ο κόσμος είναι παγιδευμένος, είναι πολιορκημένος, δεν έχει πρόσβαση ούτε σε τροφή, ούτε σε φάρμακα, ούτε στις βασικές υπηρεσίες, τα στοιχειώδη. Έχουν γίνει πρόσφατα κάποιες καταπαύσεις πυρός που ε, στο χολ, ας πούμε, σε μια γειτονιά ε, που είναι ελπιδοφόρα, αλλά δεν αρκούν. Ο στόχος ε, της καθολικής εκεχηρίας είναι επίγον οι βομβαρδισμοί σε περιοχές αμάχων, σε σχολεία και νοσοκομεία, ιδιαίτερα από το καθεστώς της Συρίας και του συμμάχους, είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό θα πρέπει παράλληλα με τις προσπάθειες που γίνονται να αρχίσει μια πολιτική διαδικασία να ζητήσουμε από όλες τις πλευρές να σταματήσουν οποιαδήποτε επίθεση ή βομβαρδισμό αμάχων στόχων ε, για να προστατεύεται ο άμαχος πληθυσμός και να γίνονται πλήρως σεβαστά όσα ορίζει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο θα ήταν όλεθρος και καταστροφή. Ενώ ελπίζουμε να αρχίσει τώρα η πολιτική διαδικασία να μην βελτιωθεί η επιτόπου κατάσταση και θα είναι τεράστια και η επίπτωση. Ε, έγινε κάποια πρόοδο στο Ιράκ στην καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους, λιγότερο όμως στη Συρία. Θα ήθελα να πω ότι η τρομοκρατική ομάδα αυτή δεν μπορεί και μάλλον δεν πρόκειται πλήρως να ιτηθεί αν συνεχιστεί ο στη Συρία. Ε, το ΝΤΑΕΣ βασίζεται ε, ε, εκεί στο χάος στη Συρία για να επιβιώσει και στο Ιράκ για να κάνει την προπαγάνδα του. Μόνο σε μια ενωμένη Συρία, μόνο σε μια Συρία που θα τερματίσει τον ίδιο της στον εμφύλιο πόλεμο και θα βρει τρόπους για τη συμφιλίωση θα καταφέρει να πατάξει διαπαντός και να εκριζώσει τον ΤΑΕΣ. Αυτές τις ημέρες και εβδομάδες που πέρασαν και ξέρω πολύ καλά αυτό που είπα ότι ισχύει δεν μπορεί κανείς μόνο να ε, πολεμάει το ΤΑΕΣ, πρέπει να το εκριζώσει. Είμαστε λοιπόν ενωμένοι και εκτός Συρίας και εντός Συρίας θα πρέπει να γίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα ήθελα καταρχάς να πω, και επιτρέψτε μου, για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο τερματισμός του πολέμου στη Συρία αφορά την ίδια μας την ασφάλεια, διότι σαφέστατα ε, είναι ε, η ήτα του ΝΤΑΕΣ και είναι και δικό μας συμφέρον. Η ομάδα υποστήριξης ε, συνεδρίασε στη Βιέννη με δύο γύρους, με δυσκολίες αλλά με επιτυχίες τελικά και μετά στη Νέα Υόρκη το Δεκέμβριο. Δύο γύροι λοιπόν που οδήγησαν σε ένα ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μάλιστα ομόφωνα το Δεκέμβριο. Και τέλος καταφέραμε να ενώσουμε τη διεθνή κοινότητα ε, σε ένα οδικό χάρτη ε, με τη, μορφή που γίνονται οι συνομιλίες στη Βιέννη για να καταλάβουν και οι Σύριοι και οι περιφερειακές δυνάμεις ότι η διεθνή κοινότητα είναι ενωμένη για να δείξει το δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί. Ζητεί το ψήφισμα ενδοσυριακές συνομιλίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Οι προετοιμασίες τώρα γίνονται αυτόν τον καιρό, όπως γνωρίζετε, και οι συνομιλίες προβλέπεται να αρχίσουν στη Γενέβη ε, καταρχήν την άλλη εβδομάδα. Το ψήφισμα ε, ορίζει και ένα εξάμεινο χρονοδιάγραμμα για να υπάρξει μια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς και αξιόπιστη και ενάμιση χρόνος για να γίνουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που να βασίζονται σε ένα Συριακό Σύνταγμα νέο. Βέβαια, όταν γίνουν αυτές οι εκλογές θα πρέπει να συμμετέχουν και οι Σύροι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός της χώρας. Στην πολιτική επίλυση ζητεί το ψήφισμα να δημιουργηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιμεχωμένων μερών και μηχανισμοί υλοποίησης και παρακολούθησης της εκεχηρίας. Όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ φιλόδοξα και το χρονοδιάγραμμα και ε, το θεματολόγιο και το πρόγραμμα. Αλλά είναι σαφές ότι εμείς δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον αυτή την κατάσταση, το status quo. Χρειάζονται υψηλοί στόχοι για να υπάρξει μια στοιχειώδη ελπίδα ότι θα αρχίσει μια διαδικασία. Όσο πλησιάζει η ειρήνη, όσο πλησιάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει μια ειρηνευτική διαδικασία και αποκτά σάρκα και οστά, βλέπουμε ότι οι αντιστάσει των εχθρών τη ειρήνης είναι πιο στεναρέ. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε την παρούσα φάση ω ένα παράθυρο ευκαιρία που δεν υπήρχε τα περασμένα έτη. Επιτρέψτε μου δεν να πω επίση ότι το παράθυρο αυτό Μπορεί να μην είναι ανοιχτό για πάντα. Αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία μπορεί να κλείσει. Και επίση θα ήθελα να τονίσω ότι πιστεύω ότι τελικά καταφέραμε να συγκεντρώσουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι για το Συριακό όλους τους διαφορετικούς περιφερειακούς παράγοντες και μεταξύ άλλων διότι καταφέραμε τον περασμένο Ιούλιο να βρούμε μια συμφωνία με το Ιράν που ανοίγει το δρόμο για ένα ενδεχόμενο, ενδεχόμενο, δεν λέω ότι είναι πραγματικότητα, ενδεχόμενο ενό διαφορετικού τύπου συνεργασίας. Θα τα πούμε αυτά στην επόμενη συζήτηση. Μ' αρέσουν τα βράδια εδώ στο κοινοβούλιο, μ' αρέσει που έρχομαι και κάθομαι πολλή ώρα, αλλά οι ε, προϋποθέσεις πληρούνται και πάλι. Θα δούμε ποιο τρόπο θα βρούμε, ο δρόμο θα είναι και δύσκολο και ανώμαλο και... Ε, προβληματικός. Ο κύριος Στέφαν Τεμιστούρα, ειδικό απεσταλμένο των ε, Ηνωμένων Εθνών, έχει την υποστήριξή μας όλων. Το θέσαμε αυτό στην ατζέντα όλων ε, των Συμβουλίων Υπουργών Εξωτερικών, ε, χθεσινό ήταν το τελευταίο, και το συζητήσαμε επί μακρόν πώς μπορούμε από κοινού να υποστηρίξουμε τη διαδικασία αυτή και το έργο του Στέφαν Τιμιστούρα. Είμαι και σε μόνιμη επικοινωνία ε, μαζί του. Πριν από λίγε μέρε τον είδα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε ακριβώς πώς θα προετοιμαστούν οι συνομιλίε και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπλακεί εκεί μαζί με τα κράτη-μέλη με συντονισμένο τρόπο για να συνεισφέρει περαιτέρω στην εφαρμογή και την υλοποίηση των ε, αποφάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Εχθέ, όπω σα είπα, οι Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν το Συριακό και εργάζονται ε, για το ψήφισμα αυτό και την εφαρμογή του. Τα κράτη-μέλη και η Ένωση θα υποστηρίξουν τις ενδοσυριακές συνομιλίες και όλη τη διαδικασία μετάβασης και ως πραγματογνωμοσύνη, δημιουργία συνένεση και διαμεσολάβηση. Υποστηρίζουμε τις εκεχηρίε και αυτή τη στιγμή ισχύσουν οι τοπικέ ε, επιμέρους και οι ε, ευρύτερε σε όλη την εθνική επικράτεια θα ε, ε, στείλουμε τη βοήθειά μας στο Συριακό λαό. Αυτό σημαίνει και ανάγκες για αποκατάσταση των υποδομών ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως προσπαθούμε να κάνουμε και στο Ιράκ. Για τις ελεύθερες περιοχές ή περιοχές όπου επικρατεί η Ρήρη και η μέσω στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξαρτήτως πρόσβασης, όπου αυτό είναι δυνατόν. Όπως γνωρίζετε είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ε, στη Συρία η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διαχείριση της Συριακής κρίσης περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν κινητοποιηθεί μέχρι τώρα. Συμφώνησαν χτες οι Υπουργοί επίσης επί μια κοινή προσέγγιση για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, την διάσκεψη του Λονδίνου για τη Συρία. Ξέρετε ότι επίκειται αυτή και η Γερμανία, το Κουβέιτ ε, και η Νορβηγία συμμετέχουν στη διοργάνωση αρχές Φεβρουαρίου στις 4 του μηνός. Ε, ουσιαστική υποστήριξη δέχεται η Τουρκία και θα συνεχίσουμε να δίνουμε πακέτα και για το Λίβανο και την Ιορδανία, όχι μόνο για να τους υποστηρίξουμε στις δικές τους προσπάθειες. Είναι αξιοθαύμαστο το έργο που κάνουν για την υποδοχή και την φιλοξενία των προσφύγων, αλλά για να ενισχύσουμε και τις αντιστάσεις των χώρων που είναι πάρα πολύ εκτεθειμένες με πάρα πολλούς τρόπους και η Ιορδανία και ο Λίβανος σε αυτή την κατάσταση. Και είμαι βεβαία ότι στη συζήτηση απόψε θα ακουστεί αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της αντοχής αυτών των δύο κρατών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μείζονες προκλήσεις που μπορεί να είναι κοινωνικές, ασφαλείας, πολιτικές, οικονομικές κτλ. Γιατί μπορεί η κρίση να γενικευθεί. Θα πρέπει επιγόντως να πάει βοήθεια εκεί σταθεροποίησης και ανθρωπιστική ε, όταν αλλάξουν τα πράγματα και το επιτρέψουν στο ιστορικό της Συρίας και αν φτάσουμε σε κάτι που να μοιάζει με ειρήνη, θα μπορέσει να αρχίσει να ανοικοδομείται η χώρα. Αργότερα, σε ένα απότερο στάδιο, ε, θα συζητήσουμε τις σημερινές εντάσεις ε, ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Εγώ έχω συζητήσει με τους Υπουργούς Εξωτερικών και των δύο Θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ε, κρίσιμο ότι οι συνομιλίες για τη Συρία προστατεύονται και δεν πρόκειται να μεταδοθούν οι εντάσει που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ιράν στην ε, Συρία, διότι τα προβλήματα είναι ήδη αρκετά έτσι. Εμεί από κοινού ω Ευρωπαίοι με ένα συντονισμένο τρόπο θα πρέπει να δρούμε και με του εταίρους μα, αρχή γενομένη από τη ΣΥΠΑ αλλά και με άλλου, για να στέλνουμε το ίδιο σαφέ μήνυμα προ όλου του συνομιλητέ στην περιοχή. Και όσοι επηρεάζουν τους μαχόμενους εντός Συρίας θα πρέπει να τους βοηθήσουν να ε, διαβούν το δύσβατο το μονοπάτι της ειρήνης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις συνομιλίες και να εγγυηθούμε ότι η διαδικασία θα είναι αξιόπιστη και θα δώσει στο Συριακό λαό τα επιθυμητά άμεσα αποτελέσματα τα όσα συμφωνήσαμε στη Βιέννη πρώτα και μετά στη Νέα Υόρκη με του διεθνεί και περιφερειακού φορεί, θα πρέπει να μεταφραστούν στην πράξη τώρα επί τόπου. Αλλιώ δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό το θέμα. Μόνο οι ΣΥΡΙ μπορούν να το κάνουν αυτό, ο λαός και τα κόμματα με τη βοήθεια τη διεθνού κοινότητα, αλλά οι ίδιοι θα πρέπει να το αναλάβουν. Η διεθνή κοινότητα είναι πρόθυμη να το κάνει. Την περασμένη εβδομάδα ε, συνείδησα ε, το συντονιστή της αντιπολίτευσης ΑΖΑΠ και ε, ε, διατράνωσα και πάλι την προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει ε, τις συνομιλίες, να δώσει ό,τι βοήθεια μπορεί και στη συνέχεια κατά τη διαδικασία της πολιτικής μετάβασης από την πρώτη στιγμή. Επίσης υποστηρίζουμε το έργο ε, του απεσταλμένου το ΟΗΕ για πλήρη συμμετοχή στις συνομιλίες όλων των πλευρών χωρίς αποκλεισμούς και τον βοηθούμε στο δύσκολο έργο του να ανοίξει το δρόμο για τις συνομιλίες αυτές. γιατί μόνο αν εκπροσωπούνται ευρέω όλες οι ομάδες στη Συρία θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη συνένεση που τόσο χρειάζεται. Θα ήθελα να πω και κάτι που συνήθως δεν αναφέρεται, αλλά ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών έχει σημασία για το πώς θα βγει η χώρα από την κρίση. Πιστεύω ότι η Συριακή κοινωνία στο εσωτερικό της χώρας θα πρωταγωνιστήσει και για την υλοποίηση και για την επαγρύπνηση κατά πόσο τηρούνται ε, οι εκεχηρίες. Υπάρχει η Συριακή κοινωνία με διάφορους τρόπους και με διάφορο, ε, διαφορετικό κάθε φορά σχήμα μπορεί να συμμετέχει και οι μητονότητες και οι θρησκευτικέ ομάδες. Δεν ε, ε, νο, νοείται ε, οποιασδήποτε ομάδας για λόγους θρησκευτικούς, εθνοτικούς κλπ. Μόνο έτσι θα προχωρήσει η συμφιλίωση και μόνο έτσι θα είναι αυτό το πιο αποτελεσματικό όπλο κατά του Νταές. Το είδαμε στο παρελθόν στο Ιράκ και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε λάθη που έγιναν εκεί σε προηγούμενα έτη. Για να δημιουργηθεί μια Συρία και να οικοδομηθεί ε, όχι θρησκευτική, δημοκρατική. Τώρα αρχίζει αυτή η προσπάθεια και η ειρήνη στη Συρία νομίζω είναι εφικτή. Το δείξαμε και πέρυσι ότι ορισμένα απίστευτα πράγματα και πολύ θετικά ε, είναι δυνατά μπορεί να ξεκινήσει η μετάβαση και μπορεί να ιτηθεί το ΝΤΑΕΣ Ισλαμικό κράτος οι διεθνείς και ε, εθνικοί ε, πρωταγωνιστές επιτέλους έχουν ενωθεί μετά από μια πενταετία πάρα πολύ οδυνηρή και πάρα πολύ μακρά. Τώρα έχει έρθει η ώρα των σύρων να δράξουν την ευκαιρία, να αρχίσουν τη μετάβαση, να τερματίσουν τον πόλεμο και να σταματήσουν τον ΤΑΕΣ. Και θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης, γιατί τους το λέμε σε όλους και προς όλους, ότι θα είμαστε στο πλευρό τους παραστάτες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε υπέρ της περιοχής η διεθνής κοινότητα για να γίνει δυνατή αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Μόλις μαθαίνω ότι κάτι σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση μπορώ να σας πω ότι η ΦΑΡΚ και η κυβέρνηση Κολομβίας ανακοίνωσαν τη συμφωνία της Αβάνας για ε, ε, κατέρωθαν κατάπαυση του πυρός και μόλις με ενημερώνει ο πρέσβης στην Πογωτά. Να το κάνουμε πιο συχνά αυτό εδώ με τη συζήτηση στην Ολομέλη. Αυτή λοιπόν ήταν μια υπέροχη είδηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Ξεκινάει λοιπόν συζήτηση για την κατάσταση στη Συρία και θα θέλαμε να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις των πολιτικών ομάδων. Γκάμπριελ, εκ μέρους του ΕΛΚ, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας, κυρία Μοκερίνη αποδείξατε ότι η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι να υπάρξει προόδος και σε πολιτικό επίπεδο και σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Να επιστήσω την προσοχή σας σε τέσσερα στοιχεία. Καταρχάς, το καταπίστευμα. Γνωρίζετε ότι για να διαχειριστούμε την ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να το κάνουμε και σήμερα και να προβλέψουμε το αύριο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, είναι μια απάντηση και στην κρίση των προσφύγων που τόσο μας απασχολεί. Είναι σαφές ότι η εξέλιξη της κατάστασης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την εμπλοκή όλων και στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης. Όχι μόνο σαν απόδειξη καλής πίστεως, αλλά έτσι ώστε να αποφύγουμε στην σύγχυση που μπορεί να δημιουργηθεί πριν από την περίοδο μετάβασης απέναντι ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Καταρχάς θα πρέπει να προσέξουμε γιατί οι διαιρέσεις ανάμεσα στην Διεθνή Ομάδα Στήριξης δεν πρέπει να δημιουργήσουν προβλήματα στις ενδοσυριακές συζητήσεις. Και δεύτερη παρατήρηση, και εδώ γνωρίζω ότι ο κ. Τεμιστούρα το το σκέφτεται αυτό είναι η συμμετοχή των γυναικών σαν επένδυση για το μέλλον. Η ανταλλαγή απόψεων που είχατε χθε επίσης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας και ο συνεχής διάλογος με το Λίβανο είναι πάρα πολύ θετικό. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης και όχι μόνο για τους ε, λόγους που επιβάλλει το προσφυγικό. Ευχαριστώ κύριος Μποστινάρο, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Θα ήθελα να πω ότι την περασμένη εβδομάδα είδαμε μια τραγωδία στη Μαντάγια Ιδού άλλη μία ε, απόδειξη της τρέλας, της παραφροσύνης που γεννάει ο πόλεμος και η βία σε μια χώρα. Βλέπουμε τα παιδιά να λιμοκτονούν στη Συρία μπροστά στα μάτια μας. Ε, επιτέλους κατάφερε να μπει ε, σε μια πολιορκημένη πόλη ανθρωπιστική ε, αυτοκινητοπομπή όπου 40.000 άνθρωποι κινδυνεύουν αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις στη Δυτική Συρία που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Μπάνκι Μου, Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, το να χρησιμοποιείς ε, ε, το λοιμό ως όπλο πολέμου είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και θα πρέπει να τιμωρείται αυστηρά. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν άμεσες ανάγκες πολιτικές. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να εφαρμοστεί το ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας και η ε, αποφάση της Βιέννης. Επίσης, ε, χρειάζεται ε, να γνωρίζουν οι πολιτικοί ότι είναι η μόνη λύση. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ειρήνη. Οι βομβαρδισμοί, μεταξύ αυτών και οι Ρώσοι, χωρίς καμία διάκριση καταστρέφουν ε, άμαχους στόχους, πολιτικούς στόχους, ε, κτίρια και ακόμα την ε, μετριοπαθή αντιπολίτευση. Όλα αυτά είναι αντιπαραγωγικά. Θα πρέπει να συμμετέχει το Ιράκ, το Ιράν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και όλοι οι γείτονε και οι τοπικοί παράγοντες σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Υπό την έννοια αυτή, καλωσορίζω και χαιρετώ τις προσπάθειες και του ΟΗΕ και τη διάσκεψη των δωρητών για τη Συρία που θα συνεδριάσει στις 4 Φεβρουαρίου. Η ειρήνη στη Συρία είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε για να εγγυηθούμε τη νίκη απέναντι στον ΤΑΕΣ και είναι και η μόνη δυνατότητα να τεθεί ένα τέρμα στις προσφυγικές ροές. Και ελπίζω η παραφροσύνη του ΤΑΕΣ αυτή να ιτηθεί. Ο κύριος Μπέλντερ για ένα λεπτό από τους συντηρητικούς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, δύο ζητήματα. Θέλω δύο ερωτήσεις ε, στη Συριακή τραγωδία. 400.000 άνθρωποι ζουν σε πολιορκημένες περιοχές. Τι γίνεται με τους χριστιανούς και με τους Κούρδους εκεί. τους ε, Η Ματάγια είναι συνώνυμο εξολόθρευσης του άμαχου πληθυσμού. Το έχουμε δει και στη Φούα, Καφράια, Λιπ, παντού σε άλλες πόλεις, στο Χαλέπι, στο Μπερεζόρ. 200.000 πολιορκούνται από το Ισλαμικό κράτος. Είναι τρομερά αυτά που ακούμε και όλες αυτές οι πόλεις ε, είναι, ε, είναι σημεία όπου πετάνε και δικά μας αεροσκάφη και τη συμμαχία. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μόνο οι Ρώσοι ρίχνουν ε, τρόφιμα και η Ευρώπη όχι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση ε, της χριστιανικής εκκλησίας ε, στις κουρδικές περιοχές. Τους κατάσχουν τα σπίτια, τις εκκλησίες, τους επιτίθενται ε, στο Άζακε και σε άλλες περιοχές χρειάζεται μια απορριπτική και κατηγορηματική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν φαίνεται. Πώς συμπεριφέρονται οι Κούρδοι στους χριστιανούς στη Συρία είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ευχαριστώ Τελίτσκα. Φιλελεύθερη δύο λεπτά. Uh, uh, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για την Κολομβία. Θα χαρώ πάρα πολύ αν μου δοθεί ευκαιρία να είμαι εδώ και μετά από δύο μήνες για να συγχαρώ τότε και για τη Συρία. Ε, πάρα πολλά από αυτά που είπατε είναι και τα δικά μου τα συμπεράσματα είναι αυτά στα οποία κατέληξα τις τελευταίες ημέρες. Αλλά επιτρέψτε μου να πω παρόλα αυτά μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, είναι σαφές ότι τα τελευταία πέντε αυτά χρόνια του πολέμου, τα χρόνια αυτά είχαν δραματικές επιπτώσεις, κυρίως επί των Συρίων, επί του άμαχου πληθυσμού, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν τις ε, ολέτριες συνέπειες ε, των ε, τρομοκρατικών επιθέσεων του Ισλαμικού κράτους στη Γαλλία, στη Ρωσία, Ρωσία, στην Τουρκία, στο Λίβανο, στη Σαουδική Αραβία. Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένε εξ αυτών. Νομίζω πέρυσι είχαμε μία έκκληση προς τους Ευρωπαίους ε, γιατί ο πόλεμος στη Συρία αναδιαμορφώνει την πολιτική σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έχουμε την απάντηση στους ε, έναντι των προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκλήθη να δραστηριοποιηθεί και τον ε, Νοέμβρη, οι επιθέσεις του Νοεμβρίου στο Παρίσι, νομίζω ότι στην πραγματικότητα οι επιθέσεις αυτές ε, συνέμεναν ότι η απειλή είναι εκείνη η οποία πλέον απασχολεί όλους τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι ε, θα επιτύχουμε στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Υπάρχουν όμως κάποιες προϋποθέσεις που θα τις διαβάσω. Πρώτον, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, Ασάτ, Ρωσία, Ιράν, θα πρέπει να δεχθούν το ψήφισμα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών και να καλύψουν κυρίως ε, το αίτημα που είναι να πάυσουν οι εμπόλεμες εχθροπραξίες, να βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη κυρίως ε, στις πολιορκούμενες περιοχές, στη Μαντάγια πρώτα απ' όλα. Η πολιτική κατάσταση δεν μπορεί να είναι εννοητή αν δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια για τους ανθρώπους στη Συρία. Δεύτερη, η προπόθεση και θα είμαι ε, πολύ θα πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή του ΦΣΑΤ και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, πρέπει να κλιμακωθούν οι προσπάθειες έτσι ώστε να γίνουν σεβαστές οι συμφωνίες οι οποίες έχουν συνομολογηθεί και τέλος αποκλιμάκωση του πολέμου στη Συρία. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του Ισλαμικού κράτους. Ε, δεν πρέπει να αποδυναμώνεται η υπόθεση της Συρίας καθώς ε, όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το Ισλαμικό κράτος εύχομαι καλή τύχη και βεβαίως είμαι ευτυχής που η τσεχική πρεσβεία στη Συρία, μία από τις τελευταίες που υπάρχουν στην περιοχή, θα σας βοηθήσουν κυρίως στην ανοικοδόμηση αλλά και στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τηρείτε υπόλοιποι το χρόνο, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και ξέρετε, μιλήσατε και σχεδόν ένα λεπτό παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Επόμενο, Επόμενος, ο κύριος Χατζηγεωργίου, παρακαλώ. Αγαπητή κυρία Μογκερίνη, δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει κανείς σε αυτή την αίθουσα που μπορεί να πει κάτι ουσιαστικό, κάτι υλοποιήσιμο για τη Συρία. Αν υπάρχει κανείς τέτοιος ανάμεσό μας, θα πρέπει να αναζητηθεί σε αυτούς σε μια χούφτα ανθρώπων μέσα σε αυτή την αίθουσα που όταν όλοι μιλούσαν για αραβική άνοιξη φωνάξαμε όσο πιο δυνατά μπορούσαμε πως έρχεται βαρύς παγωμένος αραβικός χειμώνας και τότε μας κοιτούσαν κάποιοι με θυμηδία. Σήμερα λοιπόν με τα εκατομμύρια των προσφύγων, τις εκατοντάδες χιλιάδες των νεκρών, με τους πνιγμούς στο Αιγαίο, αν υπάρχει λύση, αυτοί είναι οι ηγέτες της Ευρώπης και του κόσμου να φέρουν στο ίδιο τραπέζι τις αντιμαχόμενες πλευρές στη Συρία, φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες. Οι κίνδυνοι μεγαλώνουν με την ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν αλλά και με την πλήρη ανάπτυξη των πολεμικών μηχανών της τουρκίας κατά των κούρδων μέσα στην ίδια τη χώρα τους. αλλά για να είμαστε δίκαιοι προς όλους θέλω να σας απευθύνω μια έκκληση. κάντε ένα τηλεφώνημα κυρία μογκερίνη στον τέως πρόεδρο των ηνωμένων πολιτειών τον κύριο μπούς και πέστε του τα καθέκαστα της πολιτικής του στην περιοχή τα καθέκαστα μιας απρονοησίας και μιας πολιτικής το λέω με ηρωνία οξυδέρκειας πέστε του πέντε εκατομμύρια πρόσφυγες τριακόσιες χιλιάδες νεκροί και χιλιάδες πνιγμένοι στη μεσόγειο. απλά για να ξέρει ότι γνωρίζουμε. ευχαριστώ. And the next one, Mrs. Η κυρία Λόχμπιλερ έχει το λόγο. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Hohe Vertreterin! Die Wiener Gespräche im November hatten neue Hoffnungen auf Friedensverhandlungen in Syrien geweckt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 και μέχρι μια, έναν επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτές. Και επίσης οι Κούρδοι της ε, Συρίας θα πρέπει να συμμετάσχουν και εδώ θα πρέπει να πάρει ξεκάθαρα θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά θα πρέπει να είμαστε υπέρ μια θέση που περιλαμβάνει τους πάντες της διαπραγματεύσεις. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία καθώς και στις γειτονικές χώρες ε, στην ε, ε, συνάντηση δωρητών στο Λονδίνο το Φεβρουάριο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύσει να τεθούν στη διάθεση του πεινώντος πληθυσμού τα ανθρωπιστικά μέσα για να μην λιμοκτονήσει. Ο κύριος Μπορκέτσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στις 25 Ιανουαρίου προβλέπονται συζητήσεις όσον αφορά το ζήτημα της Συρίας. Η εκπρόσωπος θεωρεί ότι στη συνάντηση αυτή θα μπορούσαμε ενδεχομένως ε, να ζητήσουμε μία αναβολή της ε, προβλεπόμενης απόφασης γιατί δεν έχουν υπογραφεί απαραίτητες συμφωνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε ποια είναι η απαραίτητη βάση για τη συζήτηση αυτή. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι. Θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη συμφωνία. Αλλά ας δούμε και λίγο ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία. Δεν αρκεί να του καταγγέλουμε μόνο του ανθρώπου αυτού, αλλά πρέπει επίση να δούμε τι γίνεται και με την αντιπολίτευση στη Συρία, τι γίνεται με την Τουρκία, ποιο ρόλο διδραματίζει η χώρα αυτή. Ουδέποτε το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Θα ήταν επίση ενδιαφέρον να γνωρίσουμε ποια είναι η στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου από την ISIS και την πώληση των αποθεμάτων αυτών προς άλλες χώρες. Θα θέλαμε επίσης να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση στην ε, Συρία αυτή γιατί στη Συρία, στη χώρα αυτή, με συγχωρείτε, γιατί πολύ συχνά μαθαίνουμε μόνο κάποια πράγματα μέσω της Μόσχας, μέσω της Ρωσίας. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει με τις ρωσικές επιθέσεις. Να μην επαφιόμαστε μόνο στα όσα μας λέει η Ρωσία για τις επιθέσεις στη Ρωσία. Ο κύριος Κολνής έχει το λόγο. 200.000 ανθρώπινα θύματα. 300 μνημεία θησαυροί της ανθρωπότητας απειλούνται από τον Ισλαμικό βανδαλισμό. Δυστυχείς χριστιανοί εκδιώκονται, πνίγονται, στραγγαλίζονται, σκοτώνονται, σταυρώνονται. Ε, παρέ, ήμασταν μάρτυρας ε, το, αποκεφαλισμών και πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτον, να συζητήσουμε με την νόμιμη κυβέρνηση αυτής της χώρας. Ό,τι και αν νομίζουν κάποιοι. Είναι ένας συνομιλητής που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε. Δεύτερον, η Τουρκία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να σταματήσουν τη βοήθεια που δίνουν στο τζιχαντιστικό κίνημα και να συμπράξουν όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες, το Ιράν, η Ρωσία και βεβαίως τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και δεν πρέπει να έχουμε την αφέλεια να πιστεύουμε ότι θα λυθούν όλα με την εκλογική πλειοψηφία, με τη ενέργεια ελεύθερων εκλογών, στις οποίες θα συμμετάσχουν ακόμα και οι πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη χώρα και ούτω καθεξής. Οι τζιχαντιστές δεν θα δεχτούν ποτέ ε, καμία τέτοιου είδους συμφωνία. Η ειρήνη θα πρέπει να αποκατασταθεί και με την ε, δύναμη, την διεθνή δύναμη, στην οποία θα συμμετάσχουν και ε, χώρες μουσουλμανικές, όλα αυτά υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι δυτικοί βομβαρδισμοί δεν πρόκειται να φέρουν ειρήνη στη δυστυχισμένη αυτή χώρα. Ο κύριος Στετίνα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το ίσις και το καθεστώς Άσαντ είναι οι βασικοί παράγοντες, οι βασικοί δρόντες παίκτες στον εμφύλιο αυτό πόλεμο. Το καθεστώς Άσαντ όμως εξαρτάται από τους συμμάχους του. Η Ρωσία ξεκίνησε την παρέμβασή της το Σεπτέμβριο πέρσι, τη στιγμή κατά την οποία έπαιρναν το πάνω χέρι οι αντιφρονούντες σε σχέση με τον Άσαντ η Ρωσία έσωσε το καθεστώς Άσαντ και επιμήκυνε τον πόλεμο και προκάλεσε ένα νέο κύμα προσφύγων. Ορισμένες φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένες φωνές μας καλούν να συνεργαστούμε με τον Άσαντ και τους Ρώσους. Ακόμα και ο Τσέχος πρόεδρος ανοιχτά εξέφρασε τη στήραξή του στον Ασάντ. Ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τη Ρωσία για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Είναι αυτό παράλογο και σχιζοφρενικό. Δεν θα έπρεπε να το κάνουμε διότι αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστούμε με χώρες που εμπλέκονται σε κρατική τρομοκρατία. Πώς γίνεται να επιβάλλουμε κυρώσει στη Ρωσία από τη μία πλευρά και από την άλλη να συνεργαζόμαστε με εκείνη. Το καθεστώς Άσαντ είναι πολύ πιο θανατηφόρο από το ίσις. Το ίσις έχει ε, προκαλέσει 1.400 περίπου θανάτους, ενώ το καθεστώς Άσαντ πάνω από 12.000 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών. Και πολλοί Σύριοι έχουν υποστεί βασανιστήρια από το καθεστώς Άσαντ το οποίο είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, πολύ πιο επικίνδυνο από το ISIS. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος, ο κύριος Βάιντεν Χόλτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, στην Συρία διαδραματίζεται μια τρομερή καταστροφή, εκατοντάδε χιλιάδες νεκροί, κατεστραμμένο τοπίο. Το ίμιση του πληθυσμού έχει χάσει την βιωτική του βάση. Περίπου 5,5 εκατομμύρια βρίσκονται στο εξωτερικό. Όλοι γνωρίζουμε αυτούς τους αριθμούς. Οι γειτονικέ ε, περιοχές επιβαρύνονται τρομακτικά και οι ροές των προσφύγων θέτουν σε δοκιμασία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ταχύς θερματισμός του πολέμου στη Συρία είναι απολύτως αναγκαίος ε, το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών είναι το περίφημο φως στο τέλος του τούνελ ε, γιατί θέλει να συγκεντρώσει γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλους τους ενεχόμενους. Εγώ επιθυμώ κάτι να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο για τις προσπάθειές της εδώ, ε, τις οποίες ε, πολλές φορές ε, κάνει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ενώ όλοι περιμένουμε με ανεπομονησία της εξελίξεις, ο πόλεμος συνεχίζεται, οι άνθρωποι πεθαίνουν, πολλοί πεθαίνουν από την πείνα, λιμοκτονούν, οι άνθρωποι φεύγουν από το φόβο των βομβαρδισμών που έχουν σαν σκοπό να τερματίσουν ε, τον πόλεμο. Εμείς ε, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε ένα θαύμα. Χρειαζόμαστε ασφαλείς περιοχές όπου να μπορούν οι Σύροι να επιστρέψουν περισσότερο αυτό επιθυμούν. Το είδα ο ίδιος το Κομπάνι. Ε, χιλιάδες ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα του παρόλο που όλα είναι κατεστραμμένα εκεί. Ε, υπάρχουν πολλοί πολιτικοί ε, χμάλωτοι ε, πρέπει να τους ε, βαϊθήσουμε όπως τον Μπασίρ Ακταμπίλ ένας δημοκρατικός αντιφρονών δεν γνωρίζουμε κατά πόσο βρίσκεται ακόμα στη ζωή και θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο δεν είναι απαραίτητο ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την περιοχή εκεί ούτως ώστε να μπορέσουν οι Σύριοι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα που εφαρμόζεται η συμφωνία με τον Ιράν θα ήθελα να σας ε, καλέσω να ασκήσετε πίεση στο Ιράν να τερματίσει τις εχθροπραξίες στη Σύρια και να πάψει να υποστηρίζει τον Ασάντ. Τα, οι φωτογραφίες με τα παιδιά που πεθαίνουν μας υπενθυμίζουν ε, τα δεινά του πληθυσμού. Είναι 2016 και είναι σαν να έχουμε ε, ξεχάσει ότι υποσχεθήκαμε ότι δεν θα υπάρξουν ε, νέοι ε, βομβαρδισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί. Θα πρέπει πραγματικά να το απαιτήσουμε αυτό από τους ε, αυτούς μας. Ε, χωρίς τη δέσμευση της χωρίς έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα εκ μέρους της Συρίας, οι, οι, οι πρόσφυγες θα συνεχίζουν να έρχονται κατά κύματα στην Ευρώπη ε, και όλα αυτά έχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις και για την Ευρώπη τόσο η δημοκρατία του Ίσης όσο και οι ροές των προσφύγων και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν ε, περισσότερα πράγματα. Κυρία Γνωτού. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σε μερικές εβδομάδες οι Σύριοι θα γιορτάσουν μια πολύ λυπηρή επέτειο, πέντε χρόνια πολέμου. Η περίφημη αυτή αραβική άνοιξη αποτέλεσε τελικά εφιάλτη για τους λαούς στην περιοχή αυτή. Η Συρία βρίσκεται σε κατάσταση χάους. Ένα χάος όμως το οποίο έχει συμβάλει πάρα πολύ η Δύση, καθότι υποστήριξε την επανάσταση στη Συρία, την οποία υποκίνησαν πάρα πολλοί δίθεν μετριοπαθείς τζιχαντιστές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι επεμβαίνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλε δυτικέ δυνάμει, χωρί να έχουν συμβάλει όμω καθόλου. Αυτή τη στιγμή οι καθοστοτικέ δυνάμει στη Συρία κατηγορούνται για τη λιμοκτονία στη Μαντάγια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα υπάρχουν Ισλαμιστέ από την άλλη Νουστρά από άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι ε, τσιχαντιστές στην περιοχή αυτή χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται την ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία την πουλάνε σε πάρα πολύ ψηλές τιμές στη συνέχεια. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουν πληρώσει ένα πολύ ισχυρό τίμημα πάρα πολλές πόλεις, οι οποίες ε, τάχθηκαν υπέρ του καθεστώτος Ασάντ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξομαλυνθούν οι διπλωματικές μας σχέσεις με την ε, Συριακή κυβέρνηση. Επίσης, ε, η τελευταία έκθεση του Οργανισμού για την κατάργηση των χημικών ε, όπλων δείχνει, λέει συγκεκριμένα, ότι η Συριακή κυβέρνηση έχει καταστρέψει κάθε χημικό όπλο. Κύριο Κάν το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, πρόσφατα Είδαμε σκηνές φρίκης στη Μαντάγια. Η ασυτεία χρησιμοποιείται από το καθεστώς ε, Άσαντ ως όπλο πολέμου. Τρόφιμα, νερό και φάρμακα δεν μπορούν να μπαίνουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Είναι έγκλημα πολέμου. Και η Μαντάγια δεν είναι η μόνη πόλη υπό πολυερικία. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 400.000 άνθρωποι πεινούν σε 40 διαφορετικές περιοχές. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει, να υπάρχει άμεση πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Το ίσις και οι αντίστοιχοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, να αυξάνουν τη δύναμή τους για όσο χρόνο επιτρέπει η Δύση την ασυτεία, τα πασανιστήρια και τις μαζικές δολοφονίες ουσιαστικά. Πρέπει να συμφωνήσουμε επί της διαδικασίας μπορούμε να διαπραγματευτούμε, να υπάρξει πολιτική λύση. Είναι δική σας απόφαση και είναι πολύ καλή απόφαση σας κυρία Μοκερίνη, ε, για τα της Ιορδανίας. Θα πρέπει όλοι οι αντιφρονούντες να συνεργαστούν και να υπάρξει ένας ευρύ συνασπισμός μουσουλμανικών χωρών που θα καταπολεμήσει την τρομοκρατία. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλούμε τη Σαουδική Αραβία να συνεργαστούμε για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή τη κρίση, σε αυτή τη σύγκρουση και να υπάρξει ειρήνη και ευημερία για όλους στη Συρία. Έχετε μπλε κάρτα από, από, την κυρία από τον κύριο Άρνοντ. Τη δέχεστε? Ναι. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν είπε ότι το ίσις έχει ισχυρά σημεία. Συμφωνείτε μαζί του και αν ναι ποια είναι. Απάντηση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ISIS που χρησιμοποιεί το όνομα του Ισλάμ για να προκαλέσει οδύνη στον κόσμο. Πρέπει να συνεργαστούμε για να εξαλείψουμε το ISIS. Ο κύριος Κοτσολίνο παρακαλώ. Στο σημείο αυτό της βραδινής μας συζήτησης, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ενδεχομένω στην αλληλεγγύη αυτή απόψεων, είναι να σας ευχαριστήσουμε προφανώς για την πολύ σημαντική εργασία που κάνετε επί τόπου, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε ακόμα περισσότερες προσπάθειες προκειμένου οι αποφάσεις που ελήφθησαν στον ΟΗΕ και τα σχετικά ψηφίσματα που είχαμε στον ΟΗΕ το Δεκέμβριο, καθώς επίσης και ο δικός χάρτης, θα πρέπει τις επόμενες ημέρες ή τις επόμενες εβδομάδες να αποτελέσουν συγκεκριμένα πλέον μέτρα, να ελοποιηθούν. Και νομίζω ότι θα πρέπει το δικό μας το Κοινοβούλιο να σας υποστηρίξει, να εργαστούμε όλοι μαζί, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία που μας δίνεται αυτή τη στιγμή. Συντοπίω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση εν εξελίξει αυτή τη στιγμή. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, κάθε φορά που έχουμε συζητήσει εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο, ότι ουσιαστικά έχουμε μια γενιά παιδιών στη Συρία που έχει χαθεί. Μια ολόκληρη γενιά κυρίω από παιδιά, από ανήλικου. Νομίζω ότι θα πρέπει για αυτού ακριβώ να καταβληθούν πάρα πολύ σημαντικέ προσπάθειε. Και μην ξεχνάμε επίση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ανακοχή αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει όμω να έχουμε και δύο συγκεκριμένε προϋποθέσεις. Να ξεπεράσουμε αυτή τη στιγμή τη δυσπιστία που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες ομάδες που μάχονται τον Άισις και κυρίως νομίζω ότι θα πρέπει να προασπίσουμε την συμφωνία αυτή την οποία, την συμφωνία αυτή την οποία υπογράψαμε το Ιράν. Διακόπτη Πρόεδρος. Ο κύριος Φρόντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δικαιολογημένα Πεκρίνουμε το γεγονό ότι οι αποφάσει μα ή οι δηλώσεις πρόθεση της διεθνούς κοινότητα ε, ε, δεν εφαρμόζονται παρά πολύ βραδέως. Και εδώ εντάσσεται και το θέμα της Συρίας και επειδή μιλήσατε για καλέ ειδήσει που λάβατε σχέση με την Κολομβία, εγώ έχω κακέ ειδήσει. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις, γράφουν οι New York Times, Ποιο από την πλευρά τη ε, αντιπολίτευση θα κάτσει στο τραπέζι και κατά πόσο θα γίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Ε, κάθε μέρα πεθαίνουν ε, εκατοντάδες ε, ΣΥΡ γιατί όλοι επιθυμούμε την ειρήνη αλλά όλοι εφαρμόζουμε τον πόλεμο. Ε, το παράδειγμα της Μαντάγια. Ε, πώς είναι δυνατόν να φτάσαμε στο σημείο να λιμοκτονούν οι άνθρωποι. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι βεβαίως δυσχερής, αλλά έτσι όπως οι πυρηνικές διαπραγματεύσει με το Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενεργήσει πιο αποτελεσματικά, όχι μόνο λόγω των προσφύγων, αλλά και λόγω των ανθρώπων που ακόμα βρίσκονται στη ζωή στην ε, Συρία. Και ίσως θα πρέπει να ε, σταθούμε στη δουλειά και να συνενώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης, παρακαλώ. Το δράμα του Συριακού λαού συνεχίζεται με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εσωτερικούς και εξωτερικούς πρόσφυγες. Χαραμάδα ελπίδα άνοιξε μετά τις συναντήσεις της Βιέννης, όπου καταλήξαμε με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε μια καθαρή διαδικασία επίλυση. Όμω, παρά την ανθρωπιστική βοήθεια, μόλι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε πέντε νεκρού από ασυντία στην πόλη Μαντάγια, ενώ το Ντάε δολοφόνησε 135 αμάχου και απήγαγε περίπου 400. Πρέπει να αναλάβουμε πιο ενεργό ρόλο για τη συνεπή εφαρμογή του χρονοδιαγράμματο, για μια ενιαία και ειρηνική Συρία, μακριά από τα επικίνδυνα γεωστρατηγικά σενάρια που επιβολεύονται χώρε τη περιοχή. Τέλο, θέλω να αναφερθώ στο θέμα τη προσφυγική κρίση. Είναι προφανέ ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αποκλιμάκωση χωρί ομαλοποίηση στη συρία. είναι επίση απαραίτητο οι ευρωπαίοι ηγέτε να εφαρμόσουν τι αποφάσει που έχουν ληφθεί ιδιαίτερα αυτή τη μετεγκατάσταση και όχι μετά από κάθε σύνοδο γυρνώντα στι χώρε του να υπονομεύουν τη συμφωνία με την απραξία του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική λύση στη διένεξη στη Συρία. Μια πολιτική λύση που θα εμπλέκει όμως όλες τις δυνάμεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή επί τόπου. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βγούμε από τον πενταετή αυτοπόλεμο και να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη ειρήνη. Ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή που θέτει το Ισλαμικό κράτος ουσιαστικά έχει να κάνει κυρίως με την ισορροπία στην Συρία. 35 χριστιανικά χωριά αποτέλεσαν αντικείμενο επίθεσης τον, ήδη το Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ε, χάσει τη ζωή τους ή έχουν ε, αποτελέσει αντικείμενο, έχουν πέσει θύματα απαγωγής. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανεξιθρησκεία αποτέλεσε στο παρελθόν τη βάση οποιασδήποτε δημοκρατικής ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι επιτόπου να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταλήξουμε στην ειρήνη και προκειμένου να καταπολεμήσουμε το ISIS. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Μογκερίνη για όλα όσα κάνει και κυρίως για αυτό το μήνυμα ελπίδας, έστω και ισχνό που μας κομίζει σήμερα εδώ σε σχέση με το άνοιγμα ενός παράθυρου ευκαιρίας και πρέπει να το ανοίξουμε κι άλλο αυτό το παράθυρο. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να πω ότι καλό θα ήταν να εξετάσουμε περισσότερο την κατάσταση στη Συρία μετά τη σύγκρουση και έτσι θα στείλουμε και το μήνυμα στους Σύριους ακόμα και σε αυτούς που είναι στα στρατόπεδα προσφύγων ότι δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Οι χώρες αυτές δεν βοηθήθηκαν από τη Δύση, από το δημοκρατικό κομμάτι του κόσμου. Δεν τους δόθηκαν οι ανθρώπινοι πόροι για να οικοδομήσουν ένα πραγματικά δημοκρατικό Ιράκ. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα στους νέους που συνοστίζονται στις ουρές της προσφυγικές ότι η καλύτερη ελπίδα είναι να είναι έτοιμοι, να είναι καταρτισμένοι, να είναι εκπαιδευμένοι για να επιστρέψουν στη Συρία όχι μόνο για να βελτιώσουν τη δική τους ζωή αλλά για να προσφέρουν και μέλλον στον τόπο τους και πρέπει να είναι αυτό μέρος ενός νέου σχεδίου Marshall. Αυτό χρειαζόμαστε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μαρίας παρακαλώ. Ε, η ήττα του ντάεσ εξαρτάται άμεσα από το πέρας του εμφυλίου πολέμου στη συρία και τη δρομολόγηση ειρηνευτικής διαδικασίας για την πολιτική επίλυση του συριακού για δημοκρατική συγκρότηση του κράτους της συρίας νέο σύνταγμα και δημοκρατικές εκλογές. ταυτόχρονα πρέπει να απομονωθούν οι δυνάμεις που στηρίζουν και συνεργάζονται με τους τζιχαντιστέ και αυτό αφορά πρωτίστως την τουρκία τη σαουδική αραβία και το κατάρ που υποθάλπουν και βοηθούν τους τζιχαντιστές ανταυτού η ευρωπαϊκή ένωση όχι μόνο ανέχεται τα παιχνίδια της άγκυρας αλλά επιπλέον της δίνει και πρίκα τρία δισεκατομμύρια ευρώ για την εκ μέρους της τουρκίας δίθεν βοήθεια στο προσφυγικό. στο προσφυγικό όπου η τουρκία βοηθά τα δουλεμπορικά κυκλώματα που μεταφέρουν κάθε μέρα χιλιάδες πρόσφυγες στα νησιά του αιγαίου τα οποία δεν αντέχουν κυρία Μογκερίνη άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. για να γίνει λοιπόν η κατάσταση πιο ενεργητική για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα θα πρέπει τα hot spots να δημιουργηθούν εκεί που είναι οι πρόσφυγες δηλαδή να γίνουν τα hot spots στην τουρκία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν υπάρχουν ε, καθόλου εξελίξεις πρόοδοι όταν έχουμε φίλους τόσο δημοκρατικούς όσο η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία που επιτρέπουν το λαθερμπόριο όπλων και πετρελαίου. Όσον αφορά τον ε, περίφημο συνασπισμό, ο οποίος δεν έχει συντονιστεί με τις ε, κυβερνήσεις, θα πρέπει, θεωρώ, να αλλάξουμε το όραμα, την επιμονή, ε, την, τις δικές μας Θα πρέπει επίσης να, και νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε με την Συριακή κυβέρνηση το μέλλον της Συρίας δεν θα πρέπει να το καθορίσουν ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Ρωσία, αλλά οι ίδιοι οι πολίτες της ε, Συρίας. Ο κύριος Καστάλντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από τόσες αμφισημίες που ακούσαμε, είδαμε ότι έχουμε 400.000 νεκρούς, ε, πάρα πολλούς πρόσφυγες και επιτέλους φαίνεται ότι θα καταλήξουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Όλοι το θέλαμε αυτό. Πραγματικά όμω ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλέ οργανώσει, ιδίω από τη Σοδική Αραβία, που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ακραίε. Το πραγματικό όμω ερώτημα είναι το ακόλουθο. Αυτοί που πραγματικά εμπλέκονται σε αυτή τη διένεξη επιθυμούν πραγματικά την ειρήνη. Αν δούμε για παράδειγμα τη στάση τη Σαουδική Αραβία και ιδίω την ε, εκτέλεση του City Mami αμφισβητεί κανεί τελικά για το αν υπάρχει η πρόθεση αυτή. Και ποια είναι η πραγματική θέση τη Τουρκία. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε επίση τι θα γίνει με τον Μπασάρα Λασάντ. Ποια στάση θα κρατήσουμε απέναντί του. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να αποφανθούν αυτή τη στιγμή και να φέρουμε προφανώ στι Ηνωμένε Πολιτείε, στη Ρωσία και σε άλλε μεγάλε δυνάμει. Αναρωτιέμαι λοιπόν Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να μειώσουμε τους πόρους, τους οικονομικούς πόρους προς τον ΤΑΕΣ προκειμένου να έχει λιγότερα όπλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο αυτό. Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του ISIS. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι συνεχίζεται όλη αυτή η κυκλοφορία, η παράνομη κυκλοφορία πετρελαίου. Νομίζω ότι αν δεν καταφέρουμε να βάλουμε κατά της χρηματοδότησης τρομοκρατίας δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Ο κύριος Επιτίδιος έχει το λόγο κυρία Πρόεδρε. Η γνώμη μου είναι πως ε, και στην περίπτωση της Συρίας η Ευρωπαϊκή Ένωση διστάζει να εφαρμόσει την πολιτική εκείνη η οποία εγγυάται την επίλυση του προβλήματος. Απλά ασχολείται γενικά και με φιλολογικής φύσεως ενασχόληση και δεν λαμβάνει τα μέτρα εκείνα τα οποία θα επιλύσουν το πρόβλημα. Ο χρόνος επήγει, η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα κορυφώνεται καθημερινά πολλοί άμαχοι χάνουν τη ζωή τους είτε από τις συνεχιζόμενες μάχες είτε από την εγκληματική δράση του ντάεσ και η ευρωπαϊκή ένωση απλά παρατηρεί απαθώς αυτά τα οποία συμβαίνουν. είναι πολύ απλές και λίγες οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν. πρώτα απ' όλα πρέπει να απομονωθούν οι χώρες εκείνες οι οποίες ενισχύουν τους τζιχαντιστές δηλαδή τουρκία κατάρ σαουδική αραβία και δεύτερον υπό την προεδρία της ευρωπαϊκής ενώσεως πρέπει να κληθούν άμεσα σε διαπραγματεύσεις η ρωσία ο πρόεδρος ασαντ οι κούρδοι της συρίας και η συριακή αντιπολίτευση να αποφασίσουν για τη μορφή που θα έχει η νέα διακυβέρνηση της χώρας και όλοι μαζί να στραφούν εναντίον του isis να τον εξουδετερώσουν και να λήξει αυτή η επατοχυσία η οποία δεν κολακεύει την πολιτισμένη ανθρωπότητα αλλά ούτε και την ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα ότι ναι, προσπαθώ πραγματικά να δώσω κάποιες ενδείξεις, κάποια δείγματα ελπίδας, γιατί είμαι πεπισμένη ότι εάν δεν αναγνωρίσουμε τους, ε, τα σημεία ελπίδας, είναι πολύ δύσκολο να εργαστούμε για κάποια αλλαγή αλλά πράγματι ο δρόμος προς τα εκεί είναι δυσχερής και μακρύς. Και παρακαλώ μην ε, περιμένετε δραματικές ε, καμπές, ε, τουλάχιστον στο πολύ σύντομα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι είμαστε στον, να είμαστε στον ορθό δρόμο. Αλλά δυστυχώς απέχουμε πολύ από μια πύλη σειροτερματισμό του προβλήματος. Αλλά είναι αλήθεια ότι αν δούμε τι γινόταν πριν από ένα χρόνο, όταν δεν ήταν ενωμένη η ευρωπαϊκή κοινότητα και δεν υπήρξε ούτε καμία ενότητα στην περιοχή αλλά ούτε ο δικός χάρτης. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια έννοια της κατεύθυνσης προς την οποία θέλουμε να κινηθούμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, τον οδικό χάρτη, το χρονοδιάγραμμα κλπ. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ο ρόλος μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι συντονισμένη με όλες τις χώρες μέλη αυτές που κάθονται στο τραπέζι και αυτές που δεν κάθονται στο τραπέζι γιατί είναι ιδιαίτερο σημαντικό να συνεχίσουμε να θέτουμε το ζήτημα της κρίσης της Συρίας ούτως ώστε να εξασφαλίζουμε ότι και 28 χώρες μέλη συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και να εξασφαλίζουμε την πλήρη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρχει ένα συνεχές feedback. Και είμαι ε, πολύ ικανοποιημένη για την συμμετοχή και του Κοινοβουλίου που έχει πολύ ενεργό ρόλο εδώ. Θεωρώ ότι αυτό είναι ο ρόλος που μας ταιριάζει. Όχι τόσο να θέτουμε κάποιες προϋποθέσεις, αλλά να προσπαθούμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, θετικές προϋποθέσεις για μια έναρξη των συνομιλιών και να είμαστε παραγωγικοί σε στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Πολλοί από εσά θέσατε ερωτήματα σχέση με τη σύνθεση της αντιπροσωπείας ε, της αντιπολίτευσης, τον χρόνο, τους όρους, ε, τη μορφή των διαπραγματεύσεων, κατά πόσο θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα, θα καθυστερήσουν κλπ. Ε, προφανώς ε, έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο με τους υπουργού εξωτερικών, αλλά και πριν γίνει η ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα πρέπει να πω ότι Υπάρχει ωστόσο ένας συγκεκριμένος ρόλος για τον ειδικό εντεταλμένο των Ηνωμένων Εθνών που υποστηρίζεται από την ομάδα υποστηρίξης αλλά πιστεύουμε ότι και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαφυλάξουμε το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην προσπάθεια να βρεθούν οι ώρες και ο κατάλληλος χρόνος για τις διαπραγματεύσεις τις οποίες ε, τα Ηνωμένα Έθνη θα κάνουν και να εγγυθούμε ότι οι διάφοροι παράγοντες στην περιοχή αλλά και διεθνώς ε, να είναι αρκετά εξασφαλισμένοι ούτω ώστε να είναι εγγυημένος ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών. Ε, αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας τους Ευρωπαίους και θα καταστήσουμε σαφές είναι όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο ότι βρίσκονται ε, στα χέρια των Ηνωμένων Εθνών να ορίσουν ε, ακριβώ, αλλά θα πρέπει εμείς να βρούμε τρόπους να εγγυηθούμε ότι όλη η Συριακή κοινωνία, όλες οι ομάδες αυτές που παρέστησαν στο Ριάτ και αυτές που δεν παρέστησαν να συμμετάσχουν στην ε, πολιτική διαδικασία και να πολεμήσουν κατά ε, του Ισλαμικού κράτους της Αλνούσρα και των άλλων Ισλαμιστικών τρομοκρατικών ομάδων και να βρουν ε, έναν τρόπο να συμμετάσχουν σε αυτή τη ε, διαδικασία γιατί πολλοί είπαν ότι το σημείο κλειδί είναι να, οι ίδιοι οι Σύριοι να κρίνουν το μέλλον ε, της χώρας τους. Όλοι οι Σύριοι και αυτό σημαίνει όπως τόνισα και εκείνοι που βρίσκονται εκτός της Συρίας αυτή τη στιγμή. Τώρα, αυτό το οποίο είναι επίσης σημαντικό είναι κάτι το οποίο είπε ο συνάδελφος Κοτσολίνο σε σχέση με τις γενναίες των σύρων, γιατί πραγματικά έχουν απολεστεί κάποιες γενναίες σύρων, χάνουν τις ζωές τους, χάνουν τι δυνατότητες εκπαίδευσης, χάνουν την ελπίδα τους. Και αυτό είμαι υπερβολικά υψηλό, το οποίο μπορεί να στοιχίσει όχι το παρόν αλλά και δεκαετίες ε, στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά και ε, εκπαιδευτικά προγράμματα ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε μια χώρα που έχει πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευση ε, σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού να μπορέσει να συνεχίσει να επενδύει στο ίδιο τη το μέλλον. Γιατί όταν θα, πρέπει, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να εργαστούμε για την ανοικοδόμηση τη χώρα, θα πρέπει να έχουμε κάποιε γενιέ ε, σύρων οι οποίοι να είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν ενεργά στην ηλική και μη ηλική ανοικοδόμηση της χώρας, δηλαδή να έχουν τις γνώσεις, δεξιότητες, την εμπειρία, την εκπαίδευση ολόκληρων γενεών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το φροντίσουμε από τώρα. Αλλιώς θα έχουμε ε, τεράστια προβλήματα να τους βρούμε 20 ε, χρόνια μετά για παράδειγμα. Επίσης ε, να δούμε τα θέματα της ριζοσπαστικοποίησης γιατί είναι γενιές που βιώνουν μόνο την λιμοκτονία, το πόλεμο, την ζωή στα σαρτάοπεδα. Αυτοί δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθούν ως θετικοί ε, πολίτες του μέλλοντος. Ε, άρα λοιπόν ε, είναι και προς το ίδιο μας το συμφέρον να επενδύσουμε στην σταθερότητα μελλοντικά. Ε, πολλά ερωτήματα τέθηκαν σε σχέση με συζητήσεις που θα γίνουν είτε αργότερα απόψε της ε, σχέση μεταξύ Ιράν ε, και Σαδικής Αραβίας, την κατάσταση στην Τουρκία, την κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων κλπ. Θέματα τα οποία θα συζητούν σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω κάτι το οποίο είπα ήδη στο παρελθόν. Πραγματικά είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να έχω με εσά μια ανταλλαγή. Ε, είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την εργασία μου και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, ω είπατε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρότεινα ω πρώην μέλος του Κοινοβουλίου, ε, σε εθνικό επίπεδο, ε, ταπεινά θα πρότεινα να βρείτε έναν τρόπο να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να μπορεί να συστήσει σε ορισμένα θέματα κλειδιά και να μπορεί επίσης ε, να δείξει στην κοινή γνώμη ότι το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να εστιάσει σε αυτές τις βασικές ε, προτεραιότητες. Έτσι λοιπόν θα ε, πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τη δουλειά μας για να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις στα επόμενα χρόνια συνεργασίες. Κάποιος έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα για την ε, υποστήριξη της ε, Ιορδανίας σε σχέση με το εμπόριο. Ε, συζητήσαμε το θέμα αυτό με τον αρμόδιο Υπουργό και το Υπουργείο ε, Δημερός αλλά και με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων. Επίσης ε, το σύντησα με την ε, Βασίλισσα την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, στις Ιορδανίες και θα ήθελα να προτείνω να υποστηρίξουμε τη χώρα αυτή όχι μόνο οικονομικά αλλά και με, κάποιες, ε, με κάποια έκτακτα και στοχευμένα μέτρα ούτως ώστε να, διευκολυνθούν, να διευκολυνθεί το εμπόριο της Ιορδανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αναπτύσσουν κάτω από το πρίσμα της διάσκεψη στο Λονδίνο ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σε σχέση με το θέμα των προσφύγων είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί είναι πολύ σημαντική η ένταξη των Σύρων στις κοινότητες που τους υποδέχονται χωρίς ε, να, χωρίς να, προκύψουν, ε, να υπάρξουν συγκρούσεις γιατί η προοπτική φιλοξενία των Σύρων ε, προπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικές ε, συγκρούσεις και θα ήθελα να ελπίσω ότι μπορώ να υπολογίσω στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου ε, όσον αφορά και την επαρχιολική υποστήριξη για την υποδοχή των προσφύγων, για παράδειγμα στην Ιορδανία, αλλά και την έγκριση εμπορικών μέτρων που θα βοηθήσουν την Ιορδανία να επενδύσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυξη. Θα ολοκληρώσω εδώ ευχαριστώντας σας για όλες τις εισφορές σας που ήταν εξαιρετικά πολύτιμες για μένα και εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι εξελίξεις θα είναι ενθαρρυντικέ όπως ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες και θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας στην περιοχή αλλά και διεθνώς ούτε ώστε να διευκολύνουμε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία ε, που τελικά πιστεύω βρίσκεται στο σωστό, στη σωστή στοροχιά.